Ο Σόριν Μόισα εγκατέλειψε την ομάδα S&D, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, από τις 22 ε, Νοεμβρίου και ε, από τις 29 του μηνός σήμερα νίκη στην ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.